υποψήφων. Έκθεση Σικέρσκη πόσο τώρα προσαρμογή για τις ενισχύσει να αφορά το 2015. Ο κύριο Πέτερ Γιάρ. Έχετε το λόγο. Ένα λεπτό. Και καλώ του λοιπόν συναδέλφου, εφόσον δεν θέλουν να παραμένουν, να αποχωρήσουν από την αίθουσα, ώστε να μπορέσουν όσοι έχουν να κάνουν επεξήγηση ψήφου να μιλήσουν. Κύριε Γιάρ. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Δύο παρατηρήσει μόνο. Γιατί, ναι, πολύ ωραία το λένε ότι είναι μια τεχνική προσαρμογή και ε, καλούμαστε να δώσουμε το αποθεματικό ασφαλείας που είχε προβλεφθεί για τις κρίσεις. Έγινε η συζήτηση, έγινε η ψηφοφορία, αλλά υπάρχει και ένα άλλο ζήτημα στο οποίο θα ήθελα να με προσέξουν οι συνάδελφοι ότι δηλαδή πρέπει να εξασφαλίσουμε τη δυνατότητα για τη γεωργία αυτόνομα και χωρίς να χρειάζεται πολιτική υποστήριξη να ξεπερνά τις κρίσεις μόνη της. Αυτό είναι κάτι το οποίο πρέπει να απασχολήσει τις αρμόδιες επιτροπές. Άλλη μια φορά. Η καλύτερη βοήθεια είναι να μπορεί ο να βοηθήσει τον εαυτό του. Αυτό πρέπει να εξασφαλίσουμε και για τη Γεωργία. Ευχαριστώ. Σα ευχαριστώ θερμά. Ο επόμενο ομιλητή είναι ο κύριος Ντάνιελ Χάναν. Ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ω ήθιστε με αυτά τα δημοσιονομικά ζητήματα βρισκόμαστε σε τεχνικό πεδίο και συχνά λησμονούμε τις ποσότητες τα ποσά για τα οποία γίνεται λόγος, γιατί ο ανθρώπινο νου, ξέρετε, δεν είναι σχεδιασμένο για να συλλαμβάνει αυτά τα αστρονομικά ποσά. Δεν τα είχε προβλέψει η εξέλιξη. Ας προσπαθήσουμε όμως να βοηθήσουμε λίγο. Η καθαρή συμβολή του Ηνωμένου Βασιλείου ε, πέρυσι στην ευρωπαϊκό προϋπολογισμό ήταν 9,8 δισεκατομμύρια και ε, η ανάπτυξη σχετικά ήταν 19,2 δις. Θα μπορούσαμε δηλαδή να έχουμε χτίσει έως 18 νοσοκομεία του Εθνικού Συστήματος Υγείας και να έχουμε κάνει πολλά άλλα πράγματα για τους πολίτες. Αυτή λοιπόν η λιτότητα η οποία επευλήθη πρέπει να υπολογιστή. Έχουμε δαπανίσει περισσότερα από την εισφορά μας στον ευρωπαϊκό προϋπολογισμό από όσα μπορέσαμε να εξασφαλίσουμε μέσω τη περικοπής των 19,2 δισεκατομμυρίων από τον εθνικό προϋπολογισμό. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριο Ντόρμαν, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Η δανική αντιπροσωπεία αποφάσισε να μην υπερψηφίσει το σχετικό ε, ταμείο, τη σχετική αναπροσαρμογή, όσο σημαντική και αν είναι η ανάγκη για υποστήριξη, γιατί βλέπουμε ότι οι μόνοι γεωργοί οι οποίοι πληρώνουν το τίμημα της διαφωνίας και της συγκρούσεως Ευρωπαϊκής Ένωσης με τρίτες χώρες που χάνουν θέσεις εργασίας, που χάνουν δυνατότητες εξαγωγών, ήταν η γεωργοί της Δανίας. Οι άμεσες πληρωμές λοιπόν σε δανούς χρησιμοποιώντας ένα πολύ σκληρό μέτρο σε γεωργούς που ήδη υποφέρουν τα μάλα από την κρίση. Θα θέλαμε να αναζητηθούν και άλλες λύσεις, όχι μόνο πληρωμές με περιορισμένα ποσά. Και γι' αυτό καταψηφίσαμε. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρος. Η κυρία Λίδια Σέντρα Ροντρίγκε, ένα λεπτό. Ε, Ευχαριστώ, κυρία Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ του να πρικοδοτήσουμε το Ταμείο για περιπτώσεις κρίσεων που υφίστανται οι γεωργοί γιατί θεωρώ ότι είναι κάτι το πολύ σημαντικό. Πάντως θα επιφυλαχθώ να δω πώς θα αξιοποιηθεί αυτό το Ταμείο γιατί η κρίση έρχεται από κάποιες λανθασμένες αποφάσεις της Ευρωπαϊκής Ένωσης όπως ας πούμε το βέτο κατά της Ρωσίας και τώρα από την άλλη μεριά στέλνουν τα χρήματα και να δούμε πώς θα χρησιμοποιούν αυτά τα χρήματα ούτως ώστε να απαλύνουν την κατάσταση της κρίσης. Ευχαριστώ πολύ κυρία Ιβάνα Μάλετιτς ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πρόεδρε. Κάθε χρόνο κοιτάμε να δούμε πόσο πρέπει να περικοπούν οι άμεσες πληρωμές για να εξασφαλιστεί αποθεματικό κρίσος υπέρ της γεωργίας. Με βάση λοιπόν την ε, λόγο σύσταση θα έπρεπε οι αιτήσει ε, πληρωμές να μειωθούν κατά 1,9% ανά γεωργό 1,31% ανά γεωργό ε, επιλέξιμο. Εγώ πιστεύω ότι δεν πρέπει να χρησιμοποιηθεί ως επιχείρημα η κρίση ώστε οι γεωργοί να αποζημιωθούν για ζημίες που έχουν προξενήσει πολιτικές επιλογές και κρίσεις. Ιδάλλως θα πρέπει αυτό να το κάνουμε για ολόκληρο τον προπολογισμό και όχι μόνο για τη γεωργία. Όταν έχουμε να κάνουμε φυσικές καταστροφές, επιδημίες κτλ. Στη γεωργία θα χρειαστούν τα ποσά αυτά και εμείς στη γεωργία. Δεν αξιοποιούμε 100% του ποσού. Ευχαριστώ πολύ. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Μαριάννα Πέτυρ. Ένα λεπτό επίσης. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ υπερψήφισα την έκθεση για το ποσοστό προσαρμογής για τις που αφορά το 2015 για το λεγόμενο Ταμείο Κρίσεων. 4,1 εκατομμύρια ευρώ για το 2016 τον προϋπολογισμό επίσης και θεωρώ ότι τα χρήματα αυτά πρέπει να προκύψουν από τις άμεσες πληρωμές που ξεπερνούν τα 2.000 ευρώ. Η κτηνοτρόφοι μικρότερης κλίμακας θα πρέπει να προστατευτούν. Οι άλλοι θα έχουν μείωση κατά 39%. Στην Κροατία πάντως οι γεωργοί μπορούν να αξιοποιούν τα ποσά αυτά σε καταστάσεις κρίσεως. Και αυτό είναι λογικό γιατί οι Κροατοί γεωργοί δεν απορροφούν το 100% των άμεσων ενισχύσεων που προβλέπει ο Ευρωπαϊκός Προϋπολογισμός. Και έτσι η χρήση αυτού του προϋπολογισμού στο πλήρες θα λάβει χώρα μόλις το 2022 καλό την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να λάβει υπόψη και να συμπεριλάβει και να προσφέρει αποζημιώσει στου γεωργού εκείνου που έχουν υποστεί τα, περισσότερα, τα σημαντικότερα πλήγματα από το. Ε, ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Φλάνακαν για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Εγώ υποστήριξα την πρόταση γιατί θεωρώ πως πρέπει να στηριχθούν οι γεωργοί όταν αντιμετωπίζουν κρίσεις. Αυτή τη στιγμή δυστυχώ στην ε, Ιρλανδία η γεωργική πολιτική έχει μετατραπεί σε ένα θεσμικό οικοδόμημα το οποίο δημιουργεί, προξενεί την κρίση, φέρνει κρίση στη γεωργία. Στην Ιρλανδία αλλά και σε πολλές άλλες χώρες, αλλά ιδιαίτερα στην ε, Ιρλανδία βλέπουμε να ε, διαταράσσεται η ισορροπία δυνάμεων, οι μεγαλύτεροι δηλαδή γεωργοί είναι αυτοί που έχουν τις περισσότερες ενισχύσεις και οι μικρότεροι τις λιγότερες, εξού και οι μικρότεροι γεωργοί χάνουν το μεριδιό τους από την αγορά. Μόνο εκείνοι που μπορούν να έχουν μεγάλες ενισχύσεις μπορούν να λαμβάνουν δάνεια για να μπορούν να αγοράσουν τα αγροκτήματα των μικρότερης κλίμακας γεωργών. Η γεωργική λοιπόν πολιτική αντί να επιλύει την κρίση προξενεί κρίση στην Ιρλανδία ο ΔΕ Επίτροπος και τη μέλος του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος από τους α, πλούσιους γεωργούς και μέλη του ΕΛΚ της Ιρλανδίας χαρακτηρίζεται ως κομμουνιστής. Ευχαριστώ πολύ, λέει η Πρόεδρο. Τώρα περνούμε στο δεύτερο κομμάτι των επεξηγήσεων ψήφου. Πρόκειται για την έκθεση τη κυρία Νόισλ, στρατηγική τη Ευρωπαϊκή Ένωση για την ισότητα γυναικών και ανδρών μετά το 2015. Η κυρία Σόιντοροβα έχει το λόγο ω πρώτη ομιλήτρια για ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ πολύ, Πρόεδρε. Για μένα ήταν μέγα σφάλμα το ότι δεν καταφέραμε να εγκρίνουμε μία ιδιαίτερη, ιδιαίτερα περίπλοκη τροπολογία, πολύ σημαντική για την εξίσωση ανθρώπων και γυναικών, που πρότεινε μέτρα για τον ε, τρόπο με τον οποίο μπορούν οι γυναίκες να έχουν ε, πιο ισότιμη μεταχείριση στο χώρο εργασίας, καλύτερη ε, καλύτερο συγκερασμό της του επαγγελματικού με τον οικογενειακό βίο κτλ. Θα έπρεπε να, τον έχουν, να την έχουν υποστηρίξει και οι άλλες ομάδες, όχι μόνο οι δικοί μας, είμαι ότι θα πρέπει η ομάδα μας να επανέλθει στο ζήτημα αυτό και να προσπαθήσει να τροποποιήσει έτσι το κείμενο της Ευρωπαϊκής Επιτροπής. Η έκθεση της κυρίας Νόχιλ για μένα δεν μπορούσε να εγκριθεί ως εκ τούτου. Επειδή ακριβώς δεν έγιναν δεκτές οι τροπολογίες εκείνες οι οποίες θα μπορούσαν να αντισταθμίσουν τις αρνητικές ε, διατάξεις. Εκεί δηλαδή όπου είχε υπερβεί το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο τις αρμοδιότητες του. Ευχαριστώ. Ο κύριος Μάρκος Πίπερ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ δεν υπερψήφισα τον κατάλογο διεκδικήσεων για την εξίσωση ανδρών και γυναικών, παρότι είμαι υπέρ της ισότητας. Ε, ναι, είμαι υπέρ της υποστήριξης των ποσοστώσεων των γυναικών, για πιο ευέλικ, υπέρ πιο ευέλικτων μορφών εργασίας, για τις γυναίκες, είμαι κατά της βίας της βάρος των γυναικών. Πολλά όμως από τα σημαντικά θέματα που έχουν να κάνουν με την ισότητα, τα ρυθμίζουν τα κράτη-μέλη. Είναι δική τους αρμοδιότητα όταν ε, αναμειγνύεται η Ευρώπη σε ζητήματα προστασίας της μητρότητας ή όταν γίνεται λόγος σε ευρωπαϊκό επίπεδο για το δικαίωμα στην άμβλωση, παρεμβαίνουμε στα εθνικά συντάγματα των κρατών και έτσι ναι στην ισότητα, ναι στα δικαιώματα, αλλά όχι σε, αυτή, σε αυτές τις υπερβολικές εκδικήσεις εκθέσεως. Η επόμενη ομιλήτρια είναι η κυρία Τουμπράφκα Σουίτσα για ένα λεπτό. Πρόεδρε, σας ευχαριστώ πολύ ήταν πάντα στο επίκεντρο του Ευρωπαϊκού Λαϊκού Κόμματος το ζήτημα της ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών και είμαι περήφανη σήμερα ε, εδώ στην Ολομέλεια του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου που μπορώ να υπερασπίζομαι αυτές ακριβώς τις αξίες. Λυπούμε ιδιαίτερω που από την αριστερή πτέρυγα ακούστηκαν πράγματα τα οποία δεν έχουν καμία θέση στο ψήφισμα αυτό. Είχαμε προτείνει την υιοθέτηση ενό εναλλακτικού ψηφίσματο σε κάθε επίπεδο, τοπικό, περιφερειακό, εθνικό επίπεδο, σε θέματα που έχουν να κάνουν με την εκπαίδευση, με την δημόσια οικία, με τον χώρο εργασία. Είμαστε αποφασισμένοι στον αγώνα μα για την καταπολέμηση τη βία ει βάρος των γυναικών. Είμαι πεπισμένη ωστόσο ότι τον κέριο ρόλο έχουν να τον διαδραματίσουν τα κράτη-μέλη. Η Ευρωπαϊκή Ένωση δεν θα πρέπει να εμπλέκεται σε όλου αυτού του τομεί την ισότητα, ναι, την υποστηρίζουμε, αλλά πρέπει να την αντιμετωπίσουν τα κράτη-μέλη. Ορισμένοι νόμοι, επί παραδείγματι, το οικογενειακό ε, δίκαιο και ιδιαίτερα κάποια συντάγματα σε ε, επίπεδο κρατών μελών ορίζουν ζητήματα τα οποία δεν μπορούν παρά είναι θέματα α, επικουρικότητας. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Πέτερ Γιάρ για ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Πιστεύω ότι εκφράζεται ευρύτατα η πλειονοψηφία υπέρ τη ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών εδώ στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο. Είμαι πεπισμένο ότι έχουμε ακόμα πολλά να κάνουμε στην Ευρωπαϊκή Ένωση προ την κατεύθυνση αυτή. Αλλά πρέπει να διαπιστώσουμε τα εξή. Ότι έναν στόχο τέτοιο μπορούμε μόνο από κοινού, δηλαδή Ευρωπαϊκή Ένωση και κράτη-μέλη, να ε, επιτύχουμε. Και γι' αυτό είναι πολύ σημαντικό να διευθετήσουμε την τάξη των αρμοδιοτήτων και να λαμβάνει τις αρμοδιότητες ή να λαμβάνει τις αποφάσεις η Ευρωπαϊκή Ένωση μόνο εκεί όπου έχει αρμοδιότητα και να μην παρεβαίνει στους τομείς στους οποίους έχουν αρμοδιότητα τα κράτη-μέλη. Αυτό ακριβώς ήταν το κρίσιμο σημείο στην έκθεση της κυρίας Νόχιλ για, την οποία δεν μπόρεσα, για το οποίο δεν μπόρεσα να την υπερψηφίσω. Χάσαμε μια μεγάλη ευκαιρία σήμερα. Στο Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο θα μπορούσαμε να έχουμε, κάνει, να έχουμε προβεί σε μια δήλωση, σε ένα ψήφισμα με πολύ μεγάλη πλειοψηφία και λυπούμε ιδιαίτερα που δεν τα καταφέρουμε. Δεν τα καταφέραμε, σα ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Ο κύριος Δανίλ Χάνεν, ένα λεπτό. Πρόεδρε, ευχαριστώ. Όποιος ακόμη προσκολάται στην ιδέα ότι η Ευρωπαϊκή Ένωση απαρτίζει Ένωση κρατών, να κοιτάξει τον κατάλογο. Εδώ, στους καταλόγους που αφορούν αυτήν την έκθεση για την ισότητα. Δικαιώματα στην άμβλωση, διαφορέ στην αμοιβή, στον τρόπο εργασία, στι συνθήκε εργασία, στο συγκερασμό οικογενειακού και επαγγελματικού βίου. Όλα αυτά μα δείχνουν πόσο κατακαιρματισμένη είναι η εικόνα που παρουσιάζουν ε, τα ευρωπαϊκά κράτη. Καταψηφίζω φυσικά γιατί δεν θεωρώ ότι θα πρέπει να ορίζουν οι Βρυξέλλε το τι γίνεται, αλλά από την άλλη καταγγέλλω και την ε, τον εκφοβισμό με τον οποίο προσπαθούν ορισμένοι να ισχυριστούν ότι αν καταψηφίσαμε την έκθεση αυτό σημαίνει ότι δεν είμαστε υπέρ των ανθρωπίνων δικαιωμάτων και τη ισότητα των γυναικών. Όχι, το ζήτημα δεν είναι αν είμαστε υπέρ ή κατά, όλοι είμαστε υπέρ. Αλλά το ζήτημα είναι πού θα λαμβάνονται οι αποφάσει. Και τέτοιου είδου ζητήματα πρέπει να λύνονται από δημοκρατικού μηχανισμού κέντρα αποφάσεων στα κράτη-μέλη. Ακριβώ επειδή θέλουμε να ε, υπάρχει ισότητα και να εξασφαλίζονται αυτά τα δικαιώματα, θέλουμε τι αποφάσει να τι λαμβάνουν οι υπόχρεε σε λογοδοσία εθνικέ κυβερνήσει και όχι οι ανώνυμοι και μη ε, λογοδοτούντε υπάλληλοι των Βρυξελών. Ευχαριστώ. Η κυρία Χουσμένοβα. Πρόεδρε, ευχαριστώ πολύ. Υποστήριξα την έκθεση για την ισότητα μεταξύ ανδρών και γυναικών για την περίοδο μετά το 2015. Διότι πιστεύω ότι η συμπερίληψη των γυναικών στη λήψη αποφάσεων σε κάθε επίπεδο έχει τεράστια σημασία για κάθε είδους πολιτική οι μισοί πολίτες Ευρωπαϊκής Ένωσης είναι γυναίκες. Όμως αυτό δεν καταγράφεται ούτε καν στην ε, κατάρτιση των Εθνικών Κοινοβούλιων. 63,5% των βουλευτών στα Εθνικά Κοινοβούλια είναι άντρες. Γιατί, διότι τις λίστες τις εκλογικές τις ορίζουν άντρες και άρα επιλέγουν άντρες για τις εθνικές, για τις βουλευτικές εκλογές ως υποψηφίους. Γι' αυτό και ζητώ από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο να απευθύνει έκκληση προς τα Εθνικά Κοινοβούλια να επιτρέψουν στις γυναίκες να αποκτήσουν τις κατάλληλες πολιτικές που θα τις καταστήσουν ικανές να εγγραφούν σε εκλογικές λίστες και να είναι υποψήφιες. Ε, ευχαριστώ. Παύλο Ιγκλέσιας, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψηφίζουμε υπέρ της έκθεσης για την στρατηγική ισότητα ανδρών γυναικών, διότι θεωρούμε ότι έχει τη σωστή κατεύθυνση με την ευκαιρία όμως θα ήθελα να σας υπενθυμίσω, αξιότιμοι συνάδελφοι, ότι στην Ισπανία βρισκόμαστε πολύ αργά, από την, πολύ μακριά από την εκπλήρωση των στόχων της ε, ισότητας και αυτό που έχουμε είναι τις πολιτικές της λιτότητας από την Τρόικα και από τα παραδοσιακά κόμματα της χώρας που θέλουν τώρα να εκμεταλλευτούν την ανισότητα ανδρογυναικών. Θα σας το πω ξεκάθαρα έχει πρόσωπο γυναικείο η επισφαλής εργασία. Έχουν πρόσωπο γυναικείο, είναι γυναίκες αυτοί που δεν έχουν ε, αξιοπρεπή μισθό. Και ο πρώτος εχθρός της ενισότητας στην Ευρώπη και στην Ισπανία δεν είναι ο σεξισμός και ο είναι το να υποτιμούνται, να γκρεμίζονται οι κατακτήσεις των εργαζόμενων. Μάρικ Γιούρεκ, ένα λεπτό. Ευχαριστώ κυρία Πρόεδρε. Το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο πρόσφατα ενέκρινε ένα κείμενο. Αυτό το κείμενο είναι κατά ενός βασικού δικαιώματος του δικαιώματος στην ζωή. Έτσι υπονομεύεται η αξιοπιστία οποιονδήποτε δεσμευσιών μας που αφορούν τα ανθρώπινα δικαιώματα. Έτσι η Ευρώπη παίρνει ένα λάθος δρόμο. Θα πρέπει να υπάρχει συνειδητοποίηση του κόσμου στην Ευρώπη. Αλλιώ δεν θα μπορέσουμε να εξασφαλίσουμε το μέλλον τη Ευρώπη, το μέλλον του πολιτισμού. Πρόκειται για μια επιλογή μεταξύ τη ε, ζωή και αυτού το οποίο ψηφίσαμε σήμερα που είναι ο θάνατος. Η κυρία Μαριάννα Πετήρ, ένα λεπτό. Σας ευχαριστώ, Πρόεδρε. Προβληματίζομαι γιατί το Κοινοβούλιο αναλώνει τα χρήματα των φορολογουμένων ούτω ώστε να παραγάγει και να εγκρίνει κάποια τα κάποια κείμενα κατά των όσων μας ψήφισαν. Έχουμε αυτές όλες τις τροπολογίες με τις οποίες λέμε όχι στο δικαίωμα στη ζωή που έχει το κάθε ανθρωπίνο όν. Δεν βλέπω να υπάρχει διάλογος εδώ στο ημικύκλιο. Μας δίχασε βαθύτατα η έκθεση Νόχλ. Είναι αντίθετη στις βασικές μου αρχές. Γι' αυτό και την καταψήφισα. Καταψήφισα την έκθεση Νόχλ επίσης γιατί πάρα πολλές από τις διατάξεις της αντιβαίνουν στην αρχή της επικουρικότητας. 48% αυτών, 35% των διατάξεων της εκθέσεως δεν σχετίζονται με το κείμενο της έκθεσης. 42% αποτελούν δυσμενείς διακρίσεις κατά των ανδρών. Επίσης 40% περιορίζουν σημαντικά το δικαίωμα λόγου και πρόσβαση στα ΜΜΕ. Πρόκειται για κάποιου ισχυρισμού που έρχεται η έκθεση που δεν καλύπτουν, δεν έχουν επιστημονική τεκμηρίωση. Ευχαριστώ. Η κυρία Μάριαν Χάρκιν, ένα λεπτό. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Νομίζω ότι η έκθεση αυτή έχει πάρα πολλά σωστά σημεία. Αυτή την ψήφισα, όπω λέει την Πρόεδρε, θα πρέπει να καλυφθούν τα δικαιώματα των αναπήρων γυναικών, να έχουν πρόσβαση στην αγορά, να μην έχουμε ε, έχουμε μηδενική ανοχή στην ε, βία των ε, μεταξύ των δύο φίλων οπότε και θα πρέπει τα κράτη-μέλη να καταπολεμήσουν την ευάλωτη εργασία και να μην έχει πια ανθρώπινο και γυναικείο πρόσωπο η φτώχεια. για να μην έχουμε επίσης τις μηδενικές συμβάσεις αυτούς τους ορομίσθιους. Και επίσης θα πρέπει να δούμε τη διάταξη αυτή που λέει ότι θα πρέπει να μην υπάρχει ποτέ περιορισμός των αναπαραγωγικών δικαιωμάτων. Αυτά όμως περιορίζονται σχεδόν σε όλα τα κράτη-μέλη. Οπότε θα πρέπει να μην ε, έχουμε αστερομυαλιά. Οπότε εκεί δεν συμφώνησα. Ε, θα πρέπει επίσης να δούμε πώς θα έχουμε ε, στοιχεία για κάθε στατιστική που να διαχωρίζουμε με το φύλλο. Αυτό Ευχαριστώ. Ο κύριος Σον Κέλλη. Ένα λεπτό. Πρόεδρε, όπως πολλοί άλλοι συνάδελφοι που έλαβαν το λόγο τώρα και εγώ είμαι υπέρ του κειμένου για την ισότητα ανδρών γυναικών. Όμως υπάρχουν κάποιες διατάξεις του κειμένου που δεν με βρίσκουν σύμφωνο. Νομίζω ότι είναι υπερβολικές. Ψήφισα υπέρ του εναλλακτικού κειμένου του ΕΛΚ Συμφωνώ για τα θέματα τη ανισότητα, ε, τη μισθολογική, για τα θέματα τη βία μεταξύ των φίλων, αλλά θα πρέπει να κάνουμε ε, περισσότερο από αυτέ τι κατευθύνσει και θα πρέπει και μέσω τη ε, παιδεία. οι νεαροί να μάθουν ότι ποτέ δεν θα πρέπει να έχουν βία κατά κοριτσιών και γυναικών. Αν το καταφέρουμε αυτό θα είναι ένα πολύ μεγάλο πρωτοβήμα. Ευχαριστώ. Η κυρία Τζιλ Σίμουρ, ένα λεπτό επίσης. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα κατά τη Εκεί που λέει θα πει η Ευρωπαϊκή να έχει ένα υποχρεωτικό σύστημα ποσόστοσης για, το, για την εργασία. Εμείς εκλεγήκαμε χωρίς ποσόστοση και κατόπιν με ποσόστοση. Οπότε αυτό νομίζω ότι είναι πάρα πολύ μειωτικό γιατί πάρα πολλές γυναίκες δουλεύουν σκληρά σε όλη την χώρα μας ζουν σε μια μητριαρχική κοινωνία. Εκεί που ενθαρρύνονται να πετύχουν τους στόχους τους και θα πρέπει να προσέξουν όλα αυτά τα ζητήματα ε, τα οποία υπάρχουν ως φραγμή στην κοινωνία και τις εμποδίζουν να πετύχουν. Οπότε κοιτάξτε τι γίνεται με τα στατιστικά σας στοιχεία. Δεν θα πρέπει να αναγκάζεται ε, και τις εταιρείε αλλά και το κοινοβούλιο να έχουν τέτοιες υποχρεωτικές ποσοστώσεις. Thank you. Uh, next speaker is Mr. Bill Bill Etheridge, ένα λεπτό. Ευχαριστώ. Είδατε τι λέτε για την εκπαίδευση των δύο φίλων, τι, τι λέτε για την ε, οικογένεια και τι λέτε ποιος κάνει το νοικοκυριό. Μα αυτά όλα δεν είναι θέματα ούτε του κράτους, ούτε του υπερκράτους. Αυτό το ψήφισμα αποτελεί ακόμη παραπάνω ντροπή βάρος Ευρωπαϊκής Ένωσης. Είμαι περήφανος που το καταψήφισα. Όταν έρθει η μέρα του δημοψηφίσματος στο Ηνωμένο Βασίλειο, παρακαλώ και εκλυπαρώ τον λαό της χώρας μου να μην ξεγελαστεί, μην θεωρεί ότι η υπόθεση αυτή είναι εμπόριο. Όχι, όλα αυτά είναι χειραγώγηση κοινωνική και καταράγκωση των κοινωνικών αξιών. Οπότε όταν έρθει η μέρα για το δημοψήφισμα θα ψηφίσουμε την αποχώρηση και την ελευθερία. Ένα λεπτό, κύριο Κόμπερν. Κύριε Πρόεδρε, όταν προσεχώρησε στην Ευρωπαϊκή Ένωση η χώρα μου, τότε τη λέγαμε κοινή αγορά και μα λέγατε ότι πρόκειται περί εμπορική συμφωνία. Οπότε παραπλανηθήκαμε και λόγω του κόμματο UKIP και του ότι θα επιβάλλουμε το δημοψήφισμα, αυτό το σφάλμα μα θα διορθωθεί. Θα πρέπει η Ευρωπαϊκή Ένωση να αποφασίζει και να επιβάλλει την άμβλωση, ούτε την σεξουαλική διαπαιδαγώγηση στα σχολεία έναν χάρτη πορείας για τους ΛΟΑΔ ή να ε, αφιερώνονται οι πανεπιστημιακές σπουδέ και οι πανεπιστημιακοί σε κάποιο είδους ε, έρευνες για την ανισότητα των φύλων. Τι είναι αυτά, αυτά ε, πιστεύω ότι υπάρχει ελευθερία για την ομοφιλία και για τα δύο των γυναικών αλλά τελευταία ε, ασχοληθήκαμε γι' αυτό και στο ε, Σκοτσέζικο Κοινοβούλιο. Γι' αυτό και καταψήφισα αυτού του είδους την πολιτική ορθότητα, τη στρατηγική για άντρες. Αυτά είναι ανοησίες. Θα πρέπει να σας διακόψω κύριε Κόμπεν. Ο επόμενος ομιλητής είναι η κυρία Μαρία Σπυράκη και έχει ένα λεπτό. Δεν υπερψήφισα την έκθεση γιατί εκτιμώ ότι μια σειρά προβλέψεις της είναι εθνικές αρμοδιότητες. Ωστόσο, η έκθεση αυτή μπορεί να είναι μια καλή αρχή ώστε να ενθαρρυνθούν βήματα για να γεφυρωθεί το χάσμα μεταξύ ανδρών και γυναικών στην πραγματική οικονομία ξέρουμε όλοι άλλωστε το έχουμε διαβάσει ότι μόνο το πέντε των προέδρων των διοικητικών συμβουλίων στην ευρωπαϊκή ένωση είναι γυναίκες ότι μόλις το 18,6% των μελών των εποπτικών συμβουλίων είναι γυναίκες ότι μόλις το ένα τρίτο των αυτοαπασχολούμενων εκείνων που ιδρύουν επιχειρήσεις είναι γυναίκες ενώ το 60% των νέων πτυχιούχων είναι γυναίκες. τι δεν κάνουν καλά οι γυναίκες; δεν εργάζονται πολύ; δεν έχουν καινούριε ιδέες; δεν είναι συνεπείς; τα κάνουν όλα νομίζω και η παρουσία τους στην πραγματική οικονομία δεν μπορεί να διασφαλιστεί με ασφικτικές ποσοστώσεις. πρέπει να δημιουργηθεί ένα αληθινό πλαίσιο ενθάρρυνσης που θα επιτρέψει στη γυναικεία δύναμη στη γυναικεία εφευρετικότητα στη γυναικεία ευαισθησία να είναι παρούσα στην οικονομική ανάπτυξη. σας ευχαριστώ. Ευχαριστώ. Και τώρα ο κύριος Φλάνναγκαν για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης στην Ιρλανδία χιλιάδες γυναίκες εξαναγκάζονται να φύγουν με το πλοίο ή με το αεροπλάνο και να κάνουν άμβλωση στην Βρετανία. Ε, ε, μιλήσαμε για το γάμο των ομοφι... το ε, ε, ε, και ε, πολλές γυναίκες που πήγαιναν για άμβλωση στήριξαν και το γάμο των ομοφιλοφίλων. Πιστεύω ότι αν φυλάσει κανείς, αν φροντίζει παιδιά στο σπίτι, πολλές φορές δεν θεωρείται ε, αυτό εργασία. Γιατί να μην συμπεριληφθεί, να μην ε, θεωρείται ε, άνεργη μια γυναίκα η οποία φροντίζει τα παιδιά της στο σπίτι. Η μητέρα μου ε, που δεν είδε θεωρούσε τον εαυτό της άνεργο όταν φρόντιζε εμάς. Ο κύριος Βόλφ. Πολύ δεν θα ήθελα να είμαι στο, στον κατάλογο, αλλά πάντως σας ευχαριστώ. Όχι, δεν ε, έκανα τίποτε εγώ. Ε, απλώς έκανα μια χιουμοριστική παρατήρηση. Κυρία Αντιπρόεδρε, κυρίες και κύριοι, αυτή είναι μια έκθεση ίδιας πρωτοβουλίας της κυρίας Νόχη. Μια τέτοια έκθεση είναι ευκαιρία για έναν βουλευτή να παρουσιάσει ιδέες, να φτιάξει το image του και ε, δεν είναι θέμα ε, το οποίο θα απασχολήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή που θα νομοθετήσει. Ε, αυτό είναι μια ευκαιρία για ανθρώπους στην Ευρωπαϊκή Ένωση να ελέγξουν τα κράτη-έθνη στην Ευρώπη. Εγώ είμαι υπέρ της ισότητας των δύο φύλων και της, των δικαιωμάτων της γυναίκας, αλλά αυτά θα τα αποφασίσει το Βρετανικό Κοινοβούλιο και επίσης ε, ε, με το δημοψήφισμα θα έχουν την δυνατότητα οι Βρετανοί να αποφασίσουν ποιος θα ελέγχει τη ζωή τους, το, η, Ευρωπαϊκή Ένωση και η Επιτροπή ή το Βρετανικό Κοινοβούλιο. Εγώ είμαι υπέρ του Βρετανικού Κοινοβουλίου. Η... Αν η Ευρωπαϊκή Ένωση όμως ε, αποχωρήσει μετά το δημοψήφισμα, δεν θα μπορείτε να είστε εδώ και να λαμβάνετε το λόγο και αυτό θα το μετανιώσετε επίσης. Ε, και αυτό χιουμοριστικό. Τώρα, περνώ στα γερμανικά. Τώρα η έκθεση ε, Αλέσια Μαρία Μόσκα σχετικά με τα δικαιώματα διανοητικής ε, ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες. Ο κύριος Χάναν είναι εδώ. Δεν είναι εδώ πλέον. Η κυρία Ιβάνα Μάλετιτς τότε έχει το λόγο. Ευχαριστώ, Πρόεδρε. Ψήφισα υπέρ της έκθεσης για τα δικαιώματα διανοητικής ε, ιδιοκτησίας σε τρίτες χώρες. Χρειάζεται να αναλάβουμε δράση για να μειώσουμε τη ζημιά που έγινε από την ε, ε, έλλειψη των δικαιωμάτων. Οι απώλειες είναι 80 δις το χρόνο για την Ευρωπαϊκή Ένωση. Οι παραβιάσεις των δικαιωμάτων αυτών δεν αποτελούν οικονομική ζημία μόνο, αλλά αποτελούν και κίνδυνο για την υγεία των πολιτών ε, διότι πολλά φάρμακα ε, είναι απομιμήσεις. Πρέπει λοιπόν να βελτιώσουμε τα συστήματα για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας και να βοηθήσουμε τις χώρες να έχουν αποτελεσματικότερο σύστημα παρακολούθησής τους. Γι' αυτό ψήφισα υπέρ της έκθεσης. Ο επόμενος ομιλητής κανονικά θα ήταν ο κύριος Μπίλ Έθριτζ, αλλά δεν τον βλέπω στην αίθουσα. Άρα φαίνεται ότι κάποιο λάθος έγινε στον κατάλογο. Ο κύριος Γουλφ ή ο κυρίος Έθερις θα είναι λάθη το λόγο. Φαίνεται σοκηριακή πρόταση. Αύριο στο κοινοβούλιο αυτό όχι ο κύριος Έθεριτς θα λάβει το λόγο. Ευχαριστώ κύριε Αντιπρόεδρε. Αύριο στο κοινοβούλιο αυτό η συμφωνία TTIP, το πρόγραμμα εμπορίου και επενδύσεων, θα αποφασιστεί από το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο αν θα προχωρήσει δηλαδή μια συμφωνία μεταξύ Ευρωπαϊκής Ένωσης και ΕΠΑ. Επηρεάζει όλους τους πολίτες αρνητικότατα. Στη νοτιοδυτική Αγγλία ανησυχούν οι εκλογείς μου ιδιαίτερα για το ΕΣΥ. Αυτή η πρόταση ακολουθεί την ίδια κατεύθυνση. Θέλει να εξουσιοδοτήσει την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να διαπραγματευτεί στα θέματα δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας με τρίτες χώρες. Και ποιος θα ωφεληθεί από μια τέτοια συμφωνία μια μικρή ευφυής εταιρεία στο Μάντσεστερ με μια ωραία ιδέα ή οι τεράστιες πολυεθνικές που δουλεύουν σε μυστικές επιτροπές εργασίας. Ποιοι θα ωφεληθούν. Νομίζω ότι την απάντηση την ξέρετε. Και αυτός επίσης είναι ένα ακόμα λόγος ε, που συνηγορεί υπέρ της αποχώρησής μας από την Ευρωπαϊκή Ένωση. Ε, διευκρινίζω, φαίνεται ότι έγινε από την ομάδα σας το λάθος που ε, ε, διόρισε ως αγορητή τον κύριο Έθερης και όχι εσάς. Η επόμενη έκθεση είναι η έκθεση Πάβελ Σβόμποντα για το σχέδιο δράσης για τα άϊλα αγαθά. Ευχαριστώ κύριε Πρόεδρε. Ψήφισα κατά αυτού του προγράμματο δράση Αφρική που θέλει να αναθεώρησε το δικαίωμα τη πνευματική διοκτησία, διότι αυτή η έκθεση περιγράφει αυτή την μεταρρύθμιση τη οδηγία του 2001. Οι συζητήσει στην Ευρωπαϊκή, στην Επιτροπή μα των Νομικών Θεμάτων, έδειχναν ότι η σχετική αυτή διάταξη είναι κατάλληλη. Διαπιστώνουμε δε ότι η πραγματικότητα ψυχία του κόσμου δεν προσαρμόζεται στην ε, ευρωπαϊκή νομοθετική διαδικασία. Έχουμε αυτή τη μεταρρύθμιση στα πλαίσια προσπάθειας εναρμόνισης που, στην οποία είμαστε κατά και θα πρέπει να διαπιστώσουμε ότι αυτά όλα πάρα πολύ σύντομα θα είναι απειρχιωμένα. Ευχαριστώ πολύ. Ο επόμενος ομιλητής στον κατάλογο είναι ο κύριος Μόμτσιλ Νέκοφ, ο οποίος όμως δεν βρίσκεται στην αίθουσα, ούτε ο κύριος Ντάνιελ Χάναν. Δίδω λοιπόν τώρα το λόγο στην κυρία Ιβάνα Μάλετης για ένα λεπτό. Ευχαριστώ πολύ κυρία Πρόεδρε. Η οδηγία του 2004 για την επιβολή δικαιωμάτων διανοητικής διοκτησίας ήταν σημαντικό για την εναρμόνιση της νομοθεσίας διεθνώς, ώστε να υπάρχει ενιαία και ενοποιημένη προστασία των δικαιωμάτων αυτών στη μάχη, κατά της απομίμησης και προστασίας των ευρεσιτεχνιών και του copyright. Επειδή υπάρχουν πολλές παραβιάσεις ε, στο ευρωπαϊκό επίπεδο και προκαλούν μεγάλη ζημία και επειδή είναι πολύ σημαντικές οι καινοτομίες και οι νέες τεχνολογίες για την ανταγωνιστικότητα της Ευρωπαϊκής Ένωσης, υποστήριξα την έκθεση αυτή όπως και υποστήριξα τις προσπάθειες που γίνονται από την Ευρωπαϊκή Επιτροπή να ενισχύσουν περισσότερο τα δικαιώματα αυτά μέσα από ένα σχέδιο δράσης ώστε οι καινοτόμοι να μπορούν πιο εύκολα να εφαρμόζουν κανόνες σε εθνικό επίπεδο. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ πολύ. Τελευταίος ομιλητής, ο κύριος Σον Κέλλη, για ένα λεπτό. Ήταν εύκολο να αποφασίσω να ψηφίσω την έκθεση που δεν δημιουργούσε προβλήματα. Ε, στον τίτλο αναφέρεται το σχέδιο δράσης. Πολύ σημαντικό να έχεις και σχέδιο και δράση. Τα τελευταία χρόνια ε, στην Επιτροπή Ήτρα για το θέμα αυτό και συνεχώς ε, έβλεπα ε, διάφορους ε, επιχειρηματίες, μικρομεσαίες επιχειρήσεις που ανησυχούσαν για τα δικαιώματα διανοητικής ιδιοκτησίας. Αυτό είναι κάτι που πρέπει να το γνωρίζουμε, να το καταπιαστούμε και είναι σημαντικό να έχουμε και δημόσια υποστήριξη. Ε, και το κοινό να καταλάβει και να στηρίξει ε, τις προσπάθειες στο θέμα αυτό που τόσο πολύ επηρεάζουν την οικονομία, το είπε η συνάδελφος, 80 δις το χρόνο, αλλά και τη δημιουργικότητα και την ίδια τη ζωή και επιβίωση των επιχειρήσεων. Χαιρετίζω επίσης και τη δημιουργία μιας ε, ομάδας εμπειρογνωμόνων για να παρακολουθούν ε, από κοντά τις παραβιάσεις ε, σε αυτό το θέμα. Ευχαριστώ. Το τελευταίο ομιλητής. Τώρα ε, διακόπτεται η συνεδρίαση μέχρι τις 3 ε, το απόγευμα.